Pronti? Elisabeth. Elisabeth. Bene. Benvenuti a tutti, diamo inizio ai lavori. Καλώς ορίσατε όλοι. Ξεκινάμε τις εργασίες της Επιτροπής. Καταρχήν, ε, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, ε, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Όπως γνωρίζετε, στη διάρκεια του τελευταίου Συμβουλίου Υπουργών της Γεωργίας εξετάστηκαν τα προβλήματα του ελαιόλαδου. για να μπορέσει να ενημερωθεί καταλήλω η Επιτροπή μας και να μπορέσει να αποφασίσει επί τη ουσία. ζήτησε από την Εκτελεστική Επιτροπή να μας αναφέρει ε, όσα έγιναν ενώπιον τη Επιτροπή σε σχέση με αυτά τα προβλήματα και να μας πει ποια είναι τα μέτρα τα οποία εξετάζει και που θα εξεταστούν σε επόμενη διαχειριστική επιτροπή. Θα τα συζητήσουμε σήμερα στα διάφορα. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις πριν το τέλος της συνεδρίασης, τα πρακτικά θα θεωρήσουμε πως εγκρίνονται. Σας ενημερώνω ότι η σημερινή συνεδρίαση αναμεταδίδεται στο webstream. Και υπάρχει μια μικρή αλλαγή στην ημερήσια διάταξη γιατί έχουμε τους Ισπανούς συναδέλφους που έχουν καθυστερήσει κάπως λόγω ε, καθυστέρησε στις πτήσεις τους. Γι' αυτό, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ξεκινήσουμε από το σημείο 5 και μετά θα επανέλθουμε στο 4 όπου θα ψηφίσουμε. Εντάξει, ωραία, σας ευχαριστώ. Η κυρία Νεντελτσέβα είναι εδώ. Ωραία, τέλεια. Ξεκινάμε λοιπόν με το σημείο 5. Ευρωπαϊκές στατιστικές για τις μόνιμες καλλιέργειες. Η συγγήτρια είναι η Μαρία Νεντελτσέβα. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Ο κανονισμός που προτείνει η Κομισιόν έχει στόχο την ενημέρωση και την απλοποίηση του νομικού πλαισίου, του ισχύοντος νομικού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις μόνιμες καλλιέργειες. Ο κανονισμός που προτείνεται αντικαθιστά Δύο ισχύουσε νομοθετικέ πράξει. Πρόκειται για τον κανονισμό του Συμβουλίου C379 που αφορά τα, την έρευνα για τι απελοϊνικέ επιφάνειε και την 109, 129 όσον αφορά τα οποροφόρα δέντρα. Ενημερώνω ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι η 11η Απριλίου στις 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε για αυτή την έκθεση στην Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2011. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Επιτροπής που είναι εδώ και δίνω αμέσως το λόγο στην Μαρία Νεντελτσέβα ώστε να μας παρουσιάσει το σχέδιο ονομοδότησης. Μαρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι πρόκειται για νομοθετική έκθεση μετά τη θέση ισχύ τη συνθήκης της Λισαβόνας κυρίω. Οπότε εγώ ως εισηγήτρια θέλησα να ε, ευθυγραμμιστώ με τις νέες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα γεωργίας. Σε ό,τι αφορά τις μόνιμες καλλιέργειες, έδωσα έμφαση σε δύο πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μου σημεία. Το πρώτο αφορά την απλούστευση του ευρωπαϊκού πλαισίου, νομοθετικού πλαισίου για τις ε, μόνιμες καλλιέργειε και το δεύτερο σημείο είναι η κατεξουσιοδότηση πράξη. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό και προέκυψε ήδη στη συζήτηση που είχαμε πριν από μερικού μήνε στην Επιτροπή μας ήταν σε σχέση με την κατάργηση του πρώτου παραρτήματος και τη μετάθεση του περιεχομένου στο διατακτικό. Το παράρτημα 1 προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογή ε, του κανονισμού αναφέροντα τι μόνιμε καλλιέργειε για τι οποίε απαιτούνται στατιστικά στοιχεία. Κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν σημαντικό σημείο και καλό είναι να μην υπόκειται σε μεταρρύθμιση, τροπολογία ε, μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων. Γι' αυτό το περιέλαβα στο διατακτικό του, κειμένου. Σε ό,τι αφορά την απλούστευση τη ισχύουσα νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε σημαντικέ προσπάθειε για να μειώσει το γραφειοκρατικό άχθο ε, προσπαθώντα να ανταποκριθεί ταυτόχρονα σε ανάγκε τη αγορά. Έχουμε ακόμη πιο φιλόδοξη και πρότεινε κάποιε τροπολογίε προκειμένου να αποκλειστούν οι μικροκαλλιέργειε, οι λιγότερε από 0,2 εκτάρια, να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογή. Επίση, κατήργησε την ε, ταξινόμηση για τι περιφερειέ του ΝΑΤΣ 3 για ορισμένε ε, αμπελονικέ καλλιέργειε που στόχο έχουν όχι, όχι την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί δεν προβλέπεται από το ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο η ταξινόμηση με βάση τον ΝΑΤΣ 3. Μία τέτοια συμπερίληψη θα δημιουργούσε τεράστιο γραφειοκρατικό άκθο για του δικαιούχου, ενώ ούτω ή άλλω η χρήση των στατιστικών αυτών είναι αφίβολη. Σε ό,τι αφορά τη κατεξουσιαδότηση πράξη, όπω είπα από την αρχή, στόχο μου είναι να προσπίσω τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Νέα Εξουσία, επιμένοντα φυσικά στην αυστηρή εφαρμογή των αρχών που κατοχυρώνονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 για το δικαίωμα για την αρμοδιότητα των κατεξουσιοδότηση πράξεων και τη δυνατότητα εκχώρησης ε, για μία πενταετία του δικαιώματο αυτού στην Επιτροπή. Η πενταετία ξεκινάει από την ισχύ του κανονισμού. Γιατί αρχικά προτείνεται για περιόριστο διάστημα αυτή η δυνατότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε έκθεση για το θέμα αυτό το αργότερο 9 μήνες πριν τη λήξη της πενταετούς προθεσμίας και μάλιστα είναι ανανεώσιμη αυτή η πενταετία για αντίστοιχε περιόδους εκτός φυσικά και αν το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιταχθούν σε αυτή την παράταση το αργότερο τρει μήνες πριν το τέλος της κάθε προθεσμίας, της κάθε πενταετίας. Πρόκειται για αμυγός νομικά σημεία βέβαια, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είχε νόημα να εγκύψουμε ήδη από τώρα στα θέματα αυτά και να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Γιατί πολύ συχνά ε, μιλούμε τώρα τελευταία τουλάχιστον για εκτελεστικές πράξεις. Γι' αυτό και θέλω τη γνώμη των συναδέλφων για τα θέματα αυτά. Η κατεξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ εκτός και αν ε, γνωστοποιήσουν αντιρρήσεις μέσα σε ένα δίμηνο το Συμβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τη στιγμή τη κοινοποίηση ε, των καταξιοδότηση πράξεων στο Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Και η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ένα δίμηνο ακόμη με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επιμένω στα, στην προθεσμία αυτή 2 συν 2 γιατί αρχικά είχε προταθεί το 2 συν 1 για μένα είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τον δέοντα χρόνο για να αντιδράσει. Γι' αυτό τάχθηκα υπέρ του 2 2. Και μάλιστα η κατεξουδιώτηση πράξη, ή μάλλον το δικαίωμα αυτό, μπορεί να κληθεί ανα πάσα στιγμή από το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο. Και μάλιστα προσδιορίζεται ε, σε τι πράξη αφορά η ανάκληση. Και η ανάκληση αυτή ισχύει την επόμενη τη δημοσίευσή τη ε, στην επίσημη εφημερίδα ή σε μεταγενέστερη προθεσμία, εφόσον κάτι Και Μάλιστα δεν προσβάλλει την εγκυρότητα των ήδη ε, ισχυουσών ε, κατά εξουσιοδότηση πράξεων. Αυτά ως προς τα νομοθετικά σημεία και εφιστώ την προσοχή στο παράρτημα 1, στην απλούστευση και άρα την ελάφρυση του γραφειοκρατικού άκθους που ήταν πρωταρχικός μας στόχος και φάνηκε και ήδη από την πρώτη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το περασμένο φθινόπωρο και επιπλέον προσδιορίσαμε την εμβέλεια των κατεξουδότηση πράξεων και των ε, εξουσιών που εκχωρούνται στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ καλά. Ευχαριστούμε Μαρία. Εξαιρετική δουλειά και για το θέμα της ευθυγράμμισης. Γι' αυτό και θα έλεγα να ξεκινήσουμε αμέσως τη συζήτηση. Ζήτησε το λόγο η Ελίζαμπετ Γέγκλη και με ο Παπαστάμκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή ε, δουλειά στην ε, καλή έκθεση της ε, Κομισιόν. Και η Κομισιόν εδώ πέρα έχει ξεκινήσει την συζήτηση από ό,τι βλέπω και θέλει απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Ζήτησα το λόγο γιατί πέρα από τις ε, τροπολογίες της γήτριας, εγώ θα ήθελα να πάω λίγο πιο πέρα όσον αφορά την απλοποίηση, τη μείωση της γραφειοκρατίας, για να μπορέσουμε να έχουμε και κάποιες θέσεις μετά στην ε, διαπραγμάτευση. Και είχα κάνει και εγώ τότε μια έκθεση και Πράγματι είχαμε πει πως θα έπρεπε να υπάρχουν επαρκή στοιχεία αλλά να μην αναγκάζουμε κάθε φορά τους αγρότες να συλλέγουν δύο και τρεις φορές παρόμοια πράγματα. Αυτές είναι προτάσεις που θα κάνω για μια έτσι διεύρυνση. Και όσον αφορά τις μικρότερες ε, εκμεταλλεύσεις, εντάξει μπορούμε να δούμε μία αύξηση του αριθμού των ε, στρεμάτων, αλλά κατά βάση ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εργασία της. Ευχαριστώ κύριε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια, την κυρία Νετέλσεβα, για την έκθεσή της. Όπως πολύ σωστά είπε, πρόκειται για ένα νομοθετικό κείμενο και θεωρώ αριστοτεχνική ε, τη δική της παρέμβαση, τις δικές της ε, τροπολογίες σε ό,τι αφορά την ε, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θεσμικό σύστημα της ε, συνθήκης για τη λειτουργία της Ένωσης και συγκεκριμένα στις πράξεις κατηξιοδότηση βάσει του άρθρου 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ένωσης. Πολύ σημαντικό θεωρώ επίσης το γεγονός ότι η συγγήτρια προβαίνει στην αποκλειστική απαρίθμηση των καλλιεργειών, των μονίμων καλλιεργιών, μέσα στο εντός του νομοθετικού κειμένου και δεν αφήνει την ε, απαρίθμηση των μονίμων καλλιεργειών, ε, τη ρύθμιση μάλλον αυτής, στο παράρτημα. Και επομένως αυτό διασφαλίζει τη διαρκή εμπλοκή, θεσμική εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την όποια ε, τροποποίηση. Και με αυτή την έννοια βεβαίως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εδώ αυτό το, ε, το αναφέρω ε, για όλους τους συναδέλφους μας από τη στιγμή που η απαρίθμηση αυτή είναι αποκλειστική μέσα στο, σε άρθρο του, του νομοθετικού κειμένου θα πρέπει να δούμε το εύρος των μονίμων καλλιεργιών για τις οποίες, οι οποίες θα υπόκεινται στην ευρωπαϊκή στατιστική ε, αποτύπωση. Και πολύ σημαντικό θεωρώ επίσης, και τελειώνω, αυτό στο οποίο αναφέρθηκε και η, καλή, η συνάδελφος η κυρία Γέγκλε, ε, το διοικητικό βάρος των, των γεωργών για τη συγκέντρωση όλων αυτών των στατιστικών στοιχείων, τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ποιοτικά ε, με όρους ευρωπαϊκής ακρίβειας και συνέπειας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε Γιώργο. και η κυρία Ρέιμερ συζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ συγχαίρω την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Για εμένα σημαντικό είναι εδώ πέρα ο κανονισμός ε, των στατιστικών να καλύπτει μόνο επαγγελματίες ε, αγρότες. Αν είναι να πάρουμε κάθε μικρό ε, μικρή καλλιέργεια θα γίνει ένα στατιστικό χάος γιατί, γιατί θα είναι πάρα πολλά τα στοιχεία και βέβαια θα είναι και κατά προσέγγιση. Ε... Ειδικά αν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι καλλιεργούν λίγα πράγματα για να προμηθευτούν ε, για να καλύψουν οι ίδιοι τις ανάγκες τους και όχι επαγγελματικά. Για να έχουμε έτσι και μία μείωση της γραφειοκρατίας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Συγγετρία για το έργο της. Και πραγματικά έλαβε υπόψη της ευαισθησίας των αντιπροσωπιών και ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμη, γι' αυτό και φτάσαμε σε μια λύση που μας επιτρέπει τη διαπραγμάτευση προς ένα αίσιο πέρας για όλους. Σε ό,τι αφορά τα παραρτήματα 1 και 2, έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να πλουστεύσουμε ακόμη περισσότερο τα έγγραφα αυτά. Γιατί η απλούστευση αυτή θα πρέπει να είναι κάτι που θα γίνει και χάρη στο Κοινοβούλιο. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε την απλούστευση τέτοιων εγγράφων απλώς στην Κομισιόν μέσω της κατεξουσιοδότησης πράξεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να παραγωνιστεί εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό είναι αυτό που επισήμανε η κυρία Γέγκλε. Δηλαδή, ιδιαίτερα για τα αμπέλια και τις καλλιέργειες τις σχετικές, θα μπορούσαμε από, τα 0, από το 0,2 εκτάρια να φτάσουμε στα 5. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να ανεβάσουμε κάπως το κατόφλι. Ο Μάρκ Ταραμπέλα για τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ Μιλώ εξ τη ε, της ε, ομάδας μου γιατί ήμουν ασκαιώδης εισηγητής και νομίζω πως ε, η έκθεση αυτή έχει βρει το στόχο και θέλω να τη συγχαρώ για τις δύο βασικές γραμμές της έκθεσής της, αυτή που αφορά την απλοποίηση που αναφέρθηκε Ε, Νομίζω πως μπορούμε να την επιτύχουμε και ακόμα και αν ε, κάπως ε, τελειοποιήσουμε τα πράγματα μέσω των παραρτημάτων 1 και 2 παραμένει η επιτυχία αυτή και για τις κατεξοδότησες πράξεις δεν έχω αντίρρηση σε σχέση με τα όσα μας προτείνει τώρα. Επειδή ο Μιχαήλ το ανέφερε, κυρία Νεντελτσέβα, δεν ε, θέλω να σας φέρω ε, σε να απαντήσετε εσείς, αλλά πάντως είναι σαφές ότι αν η επιφάνεια είναι μικρότερη ή ίση με 0,2 εκτάρια, θα με αφήσετε να κάνω μια τροπολογία, αλλά δεν θα είναι στην κλίμακα που πρότεινε ο Μισελ Νταντέν, γιατί τότε θα αφήναμε εκτός οποιοδήποτε μικρό παραγωγό, σκέφτομαι την Ελλάδα, και άρα οι στατιστικές μας δεν θα ήταν πλήρε. Ε, αν κάνω τροπολογία θα είναι σε κάποιο μικρή κλίμακα και πάντως Είχατε την ευγένεια να κάνετε συνεδρίες και με τους κυριοδησηγητές και να μας παρουσιάσετε όλο το θέμα, δεν ήταν απλό. Εν γέννη πάντως θα ήθελα να σας, να σας χαιρετήσω για την εργασία σας και δεν έχω αντιρρήσεις. Υπάρχει μόνο αυτό το θέμα της επιφάνειας του 0,2 που θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε ελαφρώς γιατί είναι σημαντικό να μείνουμε σε μικρές επιφάνειες για να μην αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογή και από τη συλλογή των πληροφοριών τις μικρές εκμεταλλεύσεις που σε ορισμένες χώρες, επαναλαμβάνω, είναι πολυάριθμες. Bene. Ωραία. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, θα να δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Ντίας Μονιός. Το λόγο έχει ο Διευθυντής Μονιός. Και μετά θα κλείσει η κυρία Ναντελτσέβα. Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καρντόζο από Eurostat. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ αξιόλογη της έκθεση. Φαίνεται ότι πέτυχε Διάνα και το στόχο, αλλά κατανόησε και το ακολουθητέο δρόμο για την υλοποίησή του, όπως τον σκέφτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μάλιστα η συγγήτρια πρότεινε κάποιες τροπολογίες ως προς τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρκετά θετική στο μέτρο που ευθυγραμμίζονται με τους δικούς μας στόχους και τάσσονται υπέρ της απλούστευσης και της ε, διευκόλυνσης των χρηστών ως προς τη χρήση των στατιστικών στοιχείων. Υπάρχουν όμως και κάποιες ε, απλουστεύσεις που υπερβαίνουν τις αρχικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υπερβολικές αυτές απλουστεύσεις δημιουργούν περιορισμούς. Βέβαια, ο νομοθέτης είναι κυρίαρχος ως προς τη λήψη της απόφασης και μπορεί να αποφασίσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος και η ιδανικότερη λύση. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να συνεργαστεί με τα θεσμικά όργανα για την ανέβρεση μιας συμβιβαστικής λύσης που θέλουμε να είναι όσο πιο ευρία γίνεται και να διαφυλάσει τα ουσιώδη στοιχεία της πρότασής μας. Donc, euh, pour me référer à Ως προς τις επιμέρους παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών. Τώρα, θα ήθελα να πω ότι μια αισθητή αλλαγή του κατοφλίου ίσως δημιουργήσει προβλήματα. Όχι μόνο χρησιμότητας των στατιστικών στοιχείων, αλλά και συγκρισιμότητας μεταξύ των στοιχείων των κρατών μελών οι διάφορες ε, δομές των ε, καλλιεργιών, είτε είναι αυτά, αυτές αμπέλια, είτε ο, ποροφόρα, διαφέρει και από χώρα σε χώρα, αλλά και στο εσωτερικό της ίδιας χώρας. Οπότε μια ριζική αλλαγή του καταφλίου θα περιορίσει και την ε, χρησιμότητα αυτών των στοιχείων, αλλά και τη συγκρισιμότητά τους και μάλιστα όχι μόνο σε γεωγραφικό επίπεδο, αλλά και τη συγκρισιμότητα και σε χρονικό επίπεδο, σε ιστορικό επίπεδο, γιατί θα καταστεί πιο δύσκολη η σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Σε ό,τι αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξης, Εμείς προτιμούμε μια συμβαστική λύση που θα σέβεται πλήρως την ε, κοινή συμφωνία την αμοιβαία κατανόηση που είχαμε και θα εξετάσουμε τις προτάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής του Συμβουλίου συγγνώμη και του Κοινοβουλίου προκειμένου να βρούμε μία λύση που θα συνάδει και με τα προνόμια των δύο αυτών θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καρδόζο τη Eurostat και αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις από πλευράς της Κομισιόν θα δώσω το λόγο στην κυρία Νεντελτσέβα. Παρακαλώ Μαρία. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχήν όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση και θα αναφερθώ στα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω ότι ο βασικός μας στόχος είναι η μείωση του διοικητικού άχθους και από αυτό απορρέουν και οι αλλαγές που είχα προτείνει στην έκθεσή μου. Στις συζητήσεις με την Κομισιόν θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε πιο εις βάθος τη δυνατότητα να έχουμε κάποιους πίνακες ε, στα παρατήματα 2-3 σαν προαιρετικούς πίνακες, αλλά θα πρέπει αυτό να το ξανασυζητήσουμε και υπάρχει και η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι η 11η Απριλίου και είμαι ανοιχτή στι προτάσει των συναδέλφων. Δεύτερο θέμα που αναφέρθηκε αύξηση του κατοφλίου της επιφάνειας και εγώ ίδια έχω ήδη θέσει αυτή την ερώτηση να μην αυξήσουμε από το 0,2 στο 0,5 τα εκτάρια. Τώρα, πέρα από τις εξηγήσει που ακούσαμε ε, για το ποια θα είναι η χρησιμότητα αυτών των στοιχείων και η συγκρισιμότητά του, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις χώρες στις οποίες υπάρχουν λιγότερο μεγάλες επιφάνειες, πράγμα το οποίο θα έχει ως βασική αρνητική επίπτωση ότι αν αυξήσουμε το κατόφλι στο 0,5 μπορεί να φτάσει στο 10-15% της παραγωγής που δεν θα καλύπτεται. Νομίζω λοιπόν πως δεν θα ήταν σκόπιμο από πλευρά μας να αφήσουμε σε μια φαιά ζώνη ένα τέτοιο μεγάλο ποσοστό. Ήταν λοιπόν και δική μου ανησυχία αυτή και νομίζω πως το επιχείρημα που μας προτάθηκε είναι σημαντικό και γι' αυτό και σταμάτησε στο, 0,2. Όσον αφορά τι κατεξουδότηση πράξει, φυσικά και ε, φροντίζουμε για το εύρος και το πεδίο εφαρμογή και με τι εκτελεστικές πράξει, αλλά πιστεύω ότι μάλλον ε, καλά θα τα καταφέρουμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει σε καλή βάση με τη Συμβούλιο και την Επιτροπή. Είναι λεπτό το ζήτημα προφανώ, αλλά θα ήθελα να καθησυχάσω όλου του συναδέλφου που έλαβαν το λόγο ότι θα υπερασπιστώ τη θέση του Κοινοβουλίου μέχρι τέλου, αλλά μέσω συμβιβαστικών λύσεων θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια θέση νόμιμη, θεμητή και που θα μας επιτρέψει να λειτουργήσουμε, να ενεργήσουμε και στα επόμενα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Μαρία και θυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι 11 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι και η ψηφοφορία στην Επιτροπή προβλέπεται για τις 2 Μαΐου. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις μπορούμε να επανέλθουμε γιατί οι Ισπανοί συνάδελφοι κατέφθασαν στο σημείο 4 όπου πρέπει να ψηφίσουμε. Γι' αυτό να βάλετε τις κάρτες σας. Κύριε Πρόεδρε, ήρθαμε οι Ισπανοί του ΕΛΚ, αλλά ε, περιμένουμε και τους δύο σοσιαλιστές Ισπανούς. Πρέπει να φτάσουν από στιγμή σε στιγμή γιατί ήμασταν μαζί. Ναι, ναι, είναι όλα υπό έλεγχο. Ευχαριστούμε, Ρας Γκαρσία. Έφτασε και η Ράτσε. Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να σας θυμίσω το σημείο 4 αφορά την επένδυση στο μέλλον. Ένα νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μια ανταγωνιστική βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Υπεύθυνο συντάκτης ο Τζοβάνι Λαβία, επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή ή επιτροπή των δημοσιονομικών προοπτικών, η ΣΟΥΡΕ, και πρέπει να υιοθετήσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Υποβλήθηκαν 45 τροπολογίες. Τζοβάνι, θες να πάρεις το λόγο μετά την ψηφοφορία. Οπότε, αν είστε όλοι έτοιμοι... Υπάρχουν έξι ε, συμβεβαστικές τροπολογίες ε, και μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ξεκινάμε με τη συμβιβαστική 1. Συμβιβαστική 1, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία, τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. 8. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 8. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα πάμε στην συμβαστική 2. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας για τη συμβαστική 2. Εγκρίνεται. Πάμε στην ε, τροπολογία 14. Ψηφίζουμε για τη 14. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η 14 και ψηφίζουμε τώρα για τη 15. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 15. Τέλος τις ψηφοφορίες εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 τώρα. Ψηφίζουμε για τη συμβιβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Votazione aperta. Compromesso 3. Avete votato tutti su compromesso 3. Ψηφίσατε όλοι για την 3, συμβαστική 3. Ωραία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 17. Ψηφίζουμε για τη 17. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 19. 19. Ψηφίζουμε για τη 19. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 18 που ήταν χωρισμένη σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε λοιπόν για την τροπολογία 18 πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Ψηφίζουμε για τη συμβιβαστική 4. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Ψηφίζουμε για συμβιβαστική 5. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για τροπολογία 30. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την συμβιβαστική 6. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 34, Ντάντσιλα, πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε για την 34 πρώτο τμήμα. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε την ε, τροπολογία 35. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 37. 37. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Ψηφίζουμε για την 38. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την 40. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Ψηφίζουμε για τη 41. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 42. Ψηφίσατε όλοι για τη 42. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρινέται. 43. Ψηφίσατε όλοι για τη 43. Εγκρίνετε. 44. Γέγκλε. Ψηφίζουμε για τη 44. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τέλος η τροπολογία 45, Πόλσαν και άλλοι. Ψηφίζουμε για τη 45. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Ε, εγκρίνεται. Εγκρίνεται, ναι. Και τώρα ψηφίζουμε για το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Συγχαρτήρια κύριε Λαβία. Έχετε το λόγο γιατί ζητήσατε να μιλήσετε μετά από την ψηφοφορία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να παρέμβω μετά από την έγκριση της γνωμοδότησης που θα υποβάλει η δική μας Επιτροπή στην Επιτροπή Σούρε για να σας πω τα εξή. Η Επιτροπή Σούρε ήδη έχει ένα σχέδιο έκθεσης που έχει κάνει ο εισηγητής Συγκαρίγκα όπου βρίσκονται πολλά από τα πράγματα που εμείς εγκρίναμε με αυτήν την σημερινή γνωμοδότηση και ο εισηγητή τη Επιτροπή ε, ΣΟΥΡΕ είναι και έτοιμο να δεχτεί άλλε προτάσει που μπορεί να του κάνουμε σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, ο εισηγητή Γκαρίγκα είναι έτοιμος να δεχτεί ότι η χρηματοδότηση της κοινή γεωργικής πολιτικής θα παραμείνει σε ένα χωριστό τμήμα, δηλαδή σε σχέση με την πρώτη πρόταση θα τροποποιήσω ίδιο την αρχική πρόταση και θα έχουμε μια ξεχωριστή ε, ε, κεφάλαιο για την πολιτική γεωργίας και αλίας. Ε, σε σχέση με τα όσα είπε μέχρι σήμερα, ε, υπάρχουν κάποια πράγματα που ο εισηγητή δεν να, δεν είναι έτοιμο να δεχτεί και για τα οποία φαντάζομαι όσοι είναι παρόντε εδώ στην Επιτροπή, στους, όσους δηλαδή ασχολούνται με την κοινή γεωργική πολιτική, θα μπορούσαν να κάνουν μια, έναν κοινό αγώνα, γιατί κατανοώ ποιε είναι οι δυσκολίε του εισηγητή. Θα δεχτεί την δική μα πρόταση την ουσία που θέλουμε δηλαδή για την κοινή γεωργική πολιτική μετά από το 2013 πόρους τουλάχιστον ιδίου με αυτούς που προβλέπονται στο προηγούμενο πολιετές ε, πλαίσιο για το 2013 και αυτό θα το βρούμε και στην ε, πρόταση του συγητή. Όμως, δεν σκοπεύει να δεχτεί την πρόταση που ήδη έχει υποβληθεί σε αυτή την Επιτροπή νέας αξιολόγησης στο πλαίσιο των επόμενων δημοσιονομικών προϋποτικών με τη βάση του ποσοστού πληθωρισμού. Γι' αυτό σας, προ... σας ανακοινώνω πω εγώ θα υποβάλω τροπολογία και ζητώ από όλου τους φίλους ε, του γερικού προπολογισμού ανεξάρτητα από την ε, πολιτική τους απόχρωση να, το... να τη στηρίξουν για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε και μέσα στην Επιτροπή Σούρη να πετύχουμε την αναθεώρηση του κονδυλίου στο πλαίσιο της, των νέων δημοσιονομικών προοπτικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Τζοβάνι, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου. Νομίζω πω σαν ένας αγώνας ε, ολόκληρη τη επιτροπή μα. υπάρχει κάποιος που θέλει να παρέμβει. Αν όχι, ας προχωρήσουμε. Ευχαριστώ και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξης. Ευχαριστούμε, Τζοβάνι Λαβία. Σημείο 6 τροποποίηση της οδηγίας 2001 κάθετος 112 του Συμβουλίου για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ανάλογα προϊόντα που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Συντάκτρια γνωμοδότησης είναι η κυρία Βασίλικα Ντάντσιλα επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης. Η πρόταση της Επιτροπής προσπαθεί να τροποποιήσει για δεύτερη φορά την οδηγία του Συμβουλίου 2001-112 της 20 Δεκεμβρίου μάλιστα του 2001 σε σχέση με τους ε, χυμούς και ανάλογα προϊόντα προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή και να θεσπίσει κανόνες για τη σύσταση, την ονομασία τους αλλά και τους κανόνες ε, σήμανσης αυτών των προϊόντων ώστε να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της Ένωσης. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην ε, Βασιλική Ντάντζιλα που προετοίμασε τη γνωμοδότηση και που υπάρχει ήδη σε όλες τις γλώσσες και θυμίζω ότι η υποβολή τροπολογιών προβλέπεται μέχρι τις 31 Μαρτίου στις 12. Κυρία Ντάντζιλα παρακαλώ.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 lucru care ar putea duce consumatorii în eroare. Ca atare, trebuie să permitem industriei să aibă posibilitatea de a informa consumatorii că vor găsi în magazin. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ε, παραπλάνησης. Αλλά πρέπει βεβαίως να ενημερώσουμε τους ε, καταναλωτές πως δεν ε, θα υπάρχει πλέον προσθήκη ζάχαρης, αλλά δεν θα έχουν και την ένδειξη αυτή ε, Βεβαίω πρέπει να ενημερώνονται για την καταλληλότητα του φρούτου, να είναι φρέσκο, χωρίς συντηρητικά ή κάποιες διαδικασίες όπως διαδικασίες μετά την συλλογή. Όσον αφορά τους παραγωγούς πρέπει να έχουμε κατά νου πως ε, η βιομηχανία χρειάζεται λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί οπότε για να μπορέσουν όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία θα πρέπει να δώσουμε άλλους 18 μήνες για να μπορέσουν ε, να ε, πωλήσουν το στόκ το οποίο έχουν ε, συσσωρεύσει και βεβαίως αυτό είναι μεταβατικό μέτρο γιατί έχουμε ήδη προβλέψει πως τα προϊόντα που είναι ήδη στην αγορά και είχαν ετικέτες πριν από τη θέση όδη, σε ισχύ της οδηγίας μπορούν να παραμείνουν στην αγορά για 18 μήνες. Μιλάμε για 18 ε, μήνες μάξιμου μετά τη θέση ενισχύ της ε, οδηγίας. Και τέλος προτείνω στην έκθεση αυτή μετά από μία περίοδο 5 ετών κανένας παραγωγός δεν θα επιτρέπεται να γράφει στην ε, ετικέτα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Αναμένω λοιπόν τα σχόλια, της θεροπολογίες ή τις προσθήκες σας έτσι ώστε η οδηγία αυτή να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσει των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει κυρία Γιούζο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχουμε μια καλή πρόταση και μια πολύ καλή έκθεση, οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσουμε και πολλά. Και απόδειξη ο μικρός αριθμός τροπολογιών που έχουν κατατεθεί για την γνωμοδότηση. Γίνεται διαφοροποίηση εδώ μεταξύ του χυμού φρούτων και του νέκταρ ή από συμπυκνωμένο χυμό. Επίσης περιορίζεται ο αριθμό των ε, επιτρεπόμενων ε, συστατικών και μιλάει και για τις αρωματικές ουσίες. Περιλαμβάνει και το χυμό ντομάτας στο χυμό φρούτων. Είναι πολύ θετικές λοιπόν οι προτάσεις αυτές. Είναι πολύ σημαντικό όμω να ενημερώνεται ο καταναλωτής για, τις για τι διάφορε κατηγορίε και τα είδη χυμών. Γιατί οι χυμοί χωρίς ε, προσθήκη ζάχαρη πρέπει να διαφοροποιούνται από τους χυμούς με βάση συμπυκνωμένα φρούτα ή τον νέκταρ φρούτων που εκεί υπάρχει δυνατότητα προσθήκη ζάχαρης. Αυτά θα πρέπει να προσδιορίζονται για να ενημερώνεται σωστά ο καταναλωτής. Και χαίρομαι που στην πρόταση τα προσδιορίζουμε όλα αυτά. Και καλό θα ήταν να προωθήσουμε και κάποιες ενημερωτικές εκστρατείες για να ενημερωθεί ε, ο καταναλωτής για τις αλλαγές της ε, νέας αυτής της νομοθετικής πράξης. Σε ό,τι αφορά τη μεταβατική περίοδο για την αναφορά της ε, προσθήκης ζάχαρης, χωρίς την ε, υποχρεωτική, που μπορεί να αναφέρεται στους χυμούς, δίκαιο έχει συγκεκριθεί ότι αν ε, εξαφανιστεί αυτή η μία, το χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μπορεί να πανικοβληθεί ο καταναλωτής. Χρειαζόμαστε μία μεταβατική περίοδο για να προσαρμοστούν και οι παρασκευαστές, οι παραγωγοί και οι καταναλωτές. Επίσης είναι πολύ σημαντικό τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές. Αυτό το λέμε πάντα στην Επιτροπή. Θα πρέπει όλα τα προϊόντα, είτε είναι εισαγόμενα είτε είναι τοπικά και παράγονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια για την γνωμοδότησή της, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Γέγκλη. Παρακαλώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Γνωρίζουμε πως εργάζεται πάντα πάρα πολύ καλά και προσπαθεί να κάνει τα πράγματα σωστά παρόλα αυτά. Πρόταση αυτή της Κομισιόν με ανησυχεί κάπως και ως Επιτροπή Γεωργίας ε, θα δώσουμε μόνο μία γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που θα αποφασίσει εδώ πέρα συμφωνώ με την κυρία Αγιούσο. Τι γίνεται με τις εισαγόμενους συμπυκνωμένους χυμούς που πλέον δεν θα μπορούν να τους αναγνωρίσουν οι καταναλωτές. Σωστά είπε η συγγήτρια πως θα πρέπει μόνο τα καλύτερα φρούτα να χρησιμοποιούνται για τους χυμούς. Πού το ξέρουμε τι γίνεται με τα εισαγόμενα και ποιες δυνατότητες έχουμε να απαιτούμε τις ίδιες διατάξεις. Δηλαδή, με αυτά τα οποία ακούμε εδώ πέρα, τα δυσκολεύουμε πάρα πολύ τα πράγματα για εμάς. Χρειαζόμαστε, και εδώ πέρα συμφωνώ, μια μεταβατική περίοδο, γιατί ο καταναλωτής χρειάζεται χρόνο να συνηθίσει ε, σε κάτι. Και αν απαγορευτεί να γράψουμε χωρίς προσθήκη ζάχαρης, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει και μια ξεκάθαρη επισήμανση για την προέλευση και χυμών και νέκταρ. Για ολόκληρο τον ε, ευρωπαϊκό κλάδο. Άλλωστε αυτό είναι θέμα επιβίωσης. Θα πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να προσέξουμε πάρα πολύ στη διαπραγμάτευση της ε, θέσης μας. Ανιώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις στην εισηγήτρια. Πώς ε, προέκυψε αυτό το ζήτημα. Γιατί στη χώρα μου είναι μη ζήτημα. Κανείς από την περιοχή μου ή εκτός περιοχής μου δεν ήρθε σε επαφή μαζί μου γι' αυτό. Οπότε αναρωτιέμαι γιατί είναι τόσο σημαντικό. Δεύτερον, έτσι πληροφοριακά για εμένα. Βλέπω πως ε, μιλάμε εδώ πέρα για χυμούς για ανθρώπινη κατανάλωση. Ε, Προσπαθώ να σκεφτώ κάποιον χυμό φρούτου που δεν χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση. Μπορείτε να μου πληροφορήσετε αν υπάρχουν τέτοιοι. Μαρία Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγετριά μας και να της ευχαρώ γιατί παρά τα όσα ακούσαμε προηγουμένως, θεωρώ ότι το σημείο είναι πολύ σημαντικό και η γνωμοδότηση το ίδιο. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τα σχόλια της συγκήτριας. Σε ό,τι αφορά την κατάργηση της μνήας χωρίς προσθήκη ζάχαρης και της κατεξουσιοδότησης πράξης, Συστηματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τη θέση σε εφαρμογή της Συνθήκης Λισαβόνας αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Πάντως, αν καταργηθεί η μνήα χωρίς προσθήκη ζάχαρης και ζητήσουμε από τους παραγωγούς να μην περιλαμβάνουν αυτή την ετικέτα στους χυμούς τους, ίσως προβληματίσουμε τον καταναλωτή που μπορεί να προτιμήσει άλλα ποτά, άλλα αναψυκτικά ή άλλους χυμούς που θα είναι προφανές αν περιέχουν ή όχι ζάχαρη. Ενώ η χυμή φρούτων είναι πολύ υγιεινή και θρεπτική. Κρίμα λοιπόν να πληγούν από αυτή την ρύθμιση. Εγώ προτιμώ την πρόταση ηγήτρια για θέσπιση μεταβατικής περίοδου ό,τι αφορά την κατάργηση αυτής της ετικέτας, τη μία δηλαδή χωρίς προσθήκη ζάχαρη. Τώρα, για τις αρωματικές ουσίες και τη χρήση τους, νομίζω ότι η νομοθεσία μας θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την παραγωγή και να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ των χυμών και των αρωμάτων. Κάτι που δεν είναι πάντα προφανές. Σε ό,τι αφορά την κατεξουσιοδότηση πράξης, έχουν κατατεθεί τροπολογίες για τα παραρτήματα 1 και 2. Θα πρέπει να δούμε αν είναι απαραίτητες. Πάντως το θέμα των καταξιοδότηση πράξεων είναι συζητήσιμο. Ο Αντιπρόεδρος Βοητσεχόφσκι. Ευχαριστούμε και την κυρία Ταντσίλα για την πολύ ενδιαφέρουσα της γνωμοδότηση και έχω μία ερώτηση προς την εισηγητρία και ίσως και ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από ό,τι ξέρω, οι παραγωγοί χυμών χρησιμοποιούν διάφορες ε, ε, παραπλανητικές ε, διαδικασίες για να ε, παραπλανήσουν ουσιαστικά τον καταναλωτή. Γιατί αναφέρεται η φυσική γεύση του χυμού συγκεκριμένων φρούτων, αλλά μπορεί η γεύση να είναι φυσική, να μοιάζει δηλαδή με το χυμό του φρούτου, αλλά αυτό είναι παραπλανητικό, γιατί ο χυμός αυτός δεν είναι φυσικός χυμός, δεν περιλαμβάνει δεν αποτελείται μόνο από φυσικά φρούτα. Τέτοιου είδου παραπληροφόρηση πολύ συχνά τα χρησιμοποιούν οι παραγωγοί. Γι' αυτό θα πρέπει να αποφύγουμε την συμπερίληψη τέτοιων παραπλανητικών περιφερειών στην ονομασία των, προϊόν, των χυμών. Θα πρέπει όταν λέμε φυσικός χυμός είναι πραγματικά φυσικός, γιατί ε, αν υπάρχουν παραπλανητικές πληροφορίες για τη φυσική γεύση και νομίζει ο, ο καταναλωτής ότι είναι φυσικός ο χυμός, τότε αυτό πραγματικά είναι του ανταγωνισμός. Γιατί η φυσική γεύση παρόμοια με γεύση φρούτα σημαίνει ότι και ο χυμός είναι φυσικός. Αυτό θα πρέπει να αποφευθεί τέτοια παραπλάνηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέιμερς. Ευχαριστώ. Και εγώ χαιρετίζω την τοποθέτηση της ε, συναδέλφου. Καλό είναι να έχουμε αυτή τη μεταβατική περίοδο των πέντε ετών, αλλά δεν ξέρουμε πως είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μήπως μπορεί να γίνει πιο σύντομη. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό είναι πως αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πως ε, το χωρίς προσθήκη ζάχαρης έπρεπε να είναι το φυσιολογικό να μην αναφέρεται ως κάτι έξτρα και θα έπρεπε να σημαίνονται τα προϊόντα που έχουν ζάχαρη γιατί ως μητέρα ξέρω τι είναι να πηγαίνει κανείς να ψωνίζει και να προσέχει να μην μάθουν τα παιδιά στην πολύ ζάχαρη γιατί βεβαίως αυτές οι συνήθειες θα έχουν και όταν μεγαλώσουν και θα γίνουν υπέρβαρα. Οπότε θεωρώ πως η Κομισιόν είναι σε καλό δρόμο εδώ πέρα και θα ήθελα να συμφωνήσω. Ευχαριστούμε. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλο το λόγο. Δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, που είναι ο Ζεκ Ιν. από την DJ Agri. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το, την εισηγήτρια για την εξαιρετική της έκθεση. Είναι μια πρόταση σχετικά τεχνικής φύσης. Αφορά την κατανάλωση χυμών φρούτων, αλλά ταυτόχρονα είναι μια πρόταση σημαντική για τη διαφάνεια για, απέναντι στον καταναλωτή. Ε, εν γέννη, οι πρώτες προτάσεις ε, τροπολογίας είναι επικοδομητικές ε, και συγκεκριμένα η τροπολογία που επιτρέπει μια μεταβετική περίοδο για τα αποθέματα που δεν είναι ακόμα σύμμορφα με την κοινέα οδηγία στο τέλος της περίοδου μεταγραφής αυτής και θα ήθελα μόνο να υπογραμμίσω κάποιες ανησυχίες σε σχέση με τις τροπολογίες 1 και 2 για το θέμα δηλαδή της αναφοράς των προστιθέμενων ζαχάρων για να διευκρινίσουμε την σημερινή κατάσταση και την πρόθεση της Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή η χυμοί μπορεί ή όχι να περιέχουν προστιθέμενη ζάχαρη. Εν γέννη, οι χυμοί φρούτων δεν περιέχουν προστιθέμενη ζάχαρη και η σήμανση άνευ προστιθέμενη ζάχαρη, δεν εφαρμόζεται συστηματικά ακόμα και για τους χυμούς φρούτων που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, πράγμα που συμβαίνει γενικά. Με αυτή την πρόταση της Κομισιόν οι χυμοί φρούτων λοιπόν δεν θα μπορούν πλέον σε καμία περίπτωση να περιέχουν προστιθέμενα σάχαρα. Θα περιέχουν μόνο την φυσική ζάχαρη του φρούτου και άρα αυτός ο, χαρακτήρας, ο χαρακτηρισμός χωρίς προστιθέμενα ζάχαρα θα είναι πλέον ο κανόνας. Άρα λοιπόν είναι ένας κανόνας τον οποίο σίγουρα θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε στους καταναλωτές μέσα σε μια λογική προθεσμία. Και το θέμα της αναφοράς αυτής της σήμανσης είναι αμφισβητήσιμο από την νομική άποψη γιατί θα έχουμε να κάνουμε με χυμούς φρούτων που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να περιέχουν ε, ε, πρόσθετα ζάχαρα. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουν τα κράτη-μέλη μια περίοδο μεταγραφής από τη στιγμή της υιοθέτηση της οδηγίας. 18 μήνες έχουν διαθέσει τους για τη μεταγραφή και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την τροπολογία που έχει προσθεθεί και που ε, είναι επικοδομητική, δηλαδή εισαγωγή μιας μεταβατικής περίοδου για την ε, ε, κατανάλωση των αποθεμάτων που δεν θα είναι σύμμορφα με τη νέα οδηγία. Εάν δούμε την κατάσταση αυτήν την, των, των 18 μηνών, για τη διάθεση των αποθεμάτων φτάνουμε σε μια περίοδο 4 ετών στην ουσία ε, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να προσαρμοστούν αυτά τα προϊόντα. Και μετά προβλέπεται και μεγαλύτερη προθεσμία για την εξάλληψη Μάλλον, το να προδώσουμε και μεγαλύτερη προθεσμία για την εξάλληψη αυτή τη αναφορά, τη σήμανση, θα ήταν υπερβολικό. Καλύτερα είναι να γνωρίσει ο καταναλωτή εξ αρχή ε, αυτό που ισχύει και να μην ε, σηματοδοτείται κάτι το οποίο ούτω ή άλλω σέβεται τον νόμο. Εάν δηλαδή τηρηθεί η νομοθεσία, θα πρέπει να ενημερωθεί και ο καταναλωτής, αλλά όχι απαραίτητα να αναφέρεται ε, πάνω στα προϊόντα για πολύ μακρύ χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ. Ε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αυτά είχα να πω. Ε, ευχαριστούμε την Κομισιόν, τον Ζακίνη Ντάντσιλα, ε, αν θες να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσα τις προτάσεις σας με μεγάλη προσοχή. Όπως είπα, η ζάχαρη πλέον δεν προστίθεται στους χυμούς των φρούτων και να πω, ανέφερα πως δεν το ξέρουν όλοι οι καταναλωτές αυτό. Για να έχουμε λοιπόν περισσότερη διαφάνεια πρέπει να παραμείνει ε, αυτή η ετικέτα. Όσον αφορά αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βοητσεκόφσκι, πως υπάρχουν κάποιοι χυμοί που δεν ε, προέρχονται από φρούτα, αλλά από τεχνητά αρωματικά στοιχεία. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και η κυρία Γέγκλε επίσης ανέφερε την προέλευση ε, και τα φρούτα που περιέχονται στον χυμό. Έτσι πράγματι θα γίνουν τα πράγματα πολύ πιο διάφανα και θα αποφύγουμε οποιαδήποτε παραπλάνηση των καταναλωτών. Όσον αφορά την έκθεση, στόχο έχει την απλοποίηση της οδηγίας και όπως είπε η συνάδελφος η Μαρία είναι πάρα πολύ σημαντική για την υγεία μας δεδομένου του ότι 10% των μη ε, αλκοολούχων ποτών είναι χυμή και νέκταρ φρούτων. Σημείωσα λοιπόν όλες ε, τις ε, παρατηρήσεις σας, αναμένω τις τροπολογίες και ελπίζω να βρούμε μια λύση που θα ικανοποιήσει επιθυμίες των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε κυρία Ντάντσιλα και Περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι το 7. Τροποποίηση του κανονισμού ΕΚ 378-2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την εφαρμογή της προαιρετικής διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ε, η συγκήτρια είναι η κυρία Ρέιμερς. Έκθεση του σχεδίου, ε, εξέταση συγγνώμη, του σχεδίου έκθεσης. Έχουμε να κάνουμε ευθυγράμμιση στη Λισαβόνα. Πρόταση τροποποίηση λοιπόν του κανονισμού για να ευθυγραμμιστεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η εισαγήτρια στηρίζει την χρήση της συνθήκης της ε, Λισαβόνας ε, για τις, για τις εκτελεστικές πράξεις. Κυρία Ρέιμερς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την ε, ευθυγράμμιση προς διατάξεις της ε, Συνθήκης Λισαβόνας υπάρχει η δυνατότητα μιας ε, διάρθρωσης και βεβαίως αυτό δημιουργεί προβλήματα στα κράτη-μέλη όσον αφορά τις πληρωμές κοινή ε, γεωργικής πολιτικής. Είναι πάρα πολύ τεχνική έκθεση, αφορά την διαδικασία. Η πρόταση της ε, Κομισιόν είναι να μιλήσουμε για εφαρμοστικές ε, πράξεις και μετά την προσαρμογή αυτή έχουμε γενικές αρχές όπως χρήση σε περιφερειακό επίπεδο, τα δε κράτη-μέλη σύμφωνα με το άρθρο 291 της, ε, της συνθήκης είναι υπεύθυνα για θέσεις κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανικούς ελέγχους. Θέλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε αυτή την ε, προαιρετική διάρθρωση. Βεβαίως ένα κράτος μέλος, η Μεγάλη Βρετανία, χρησιμοποιεί κάτι τέτοιο και η Πορτογαλία αποχώρησε πρόσφατα από αυτή τη διαδικασία, οπότε μόνο ένας ε, κράτος μέλος θα χρησιμοποιεί αυτή τη διαδικασία μέχρι την επόμενη μεταρρύθμιση, οπότε δεν βλέπω προβλήματα εδώ πέρα μέχρι με την πρώτη Κομισιόν να μένουμε τροπολογίες μέχρι τις 12 Απριλίου και θα τις επεξεργαστούμε. Ευχαριστώ. 12... Ευχαριστούμε. Τροπολογίες λοιπόν 12 Απριλίου 2011 στις 12. Εάν δεν υπάρχει κανείς που να θέλει να πάρει το λόγο, να δώσω αμέσω το λόγο στην ε, Σούζα Ούβα, που είναι εκπρόσωπος της Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Voilà. Merci bien, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έρχομαι στην Επιτροπή σας, ε, την Επιτροπή Γεωργίας, όπως πάντα, και μάλιστα για μια πρόταση που όπως ακούσαμε δεν είναι καθόλου αμφιλεγόμενη. Γιατί με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώσαμε ότι η της έκθεσης ε, συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ε, ακούσατε, πρόκειται για μια πρόταση ευθυγράμμισης. Η πρόταση αυτή αφορά ένα και μόνο κράτο μέλος, το Ηνωμένο Βασίλειο. Και μόνο για μία χρονιά, το 2012. Και μια και η Πορτογαλία αρνήθηκε την προαιρετική διαφοροποίηση, έχουμε αυτή την πρόταση. Η πρόταση δεν απάδει από το status quo και αν έχουμε ένα πλήρη status quo, αν έχουμε προσδιορισμό των ποσών η πρόταση προβλέπει ότι ο προσδιορισμός των ποσών ήδη έχει γίνει. Μία αλλαγή γίνεται του προσδιορισμένου ποσού. Και αυτό οφείλουμε να επιστρέψουμε το ποσό που έχει προκαταβάλει το κράτος μέλος. Και αυτό γίνεται χωρίς ε, καμία επέμβαση της Επιτροπής. Αν πρόκειται όμως για δημοσιονομική πειθαρχία ή για ε, κανονιστική ρύθμιση που σχετίζεται με την προαιρετική διαφοροποίηση στα πλαίσια του κανονισμού της αγροτικής ανάπτυξης, τότε στις δύο αυτές περιπτώσεις, που είναι μάλλον υποθετικές και απίθανες, τότε ισχύει η εκτελεστική διαδικασία. Γι' αυτό και χρειάζεται η γνωμοδότηση της ε, Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε αυτή την περίπτωση που δεν έχει αλλάξει τίποτα και μόνο αν υπάρξει κάποια αλλαγή σε σχέση με το ποσό αυτό που είναι προσδιορισμένο το πεδίο εφαρμογή αφορά μόνο μία χρονιά και μόνο μία χώρα, το 2010 και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε, δεν συμφωνούμε με τι τροπολογίε 1 και 3. Γιατί αυτέ οι δύο τροπολογίε προτείνουν τη διαδικασία της επιτροπολογίας για τον προσδιορισμό των ποσών. Μόνο αυτές τις δύο τροπολογίες διαφωνούμε. Οι υπόλοιπε είναι συντακτικής φύσης και δεν μας ε, προβληματίζουν. Οι τροπολογίες 2, 4 και 5 δηλαδή δεν είναι καθόλου αμφιλεγόμενες. Αυτά προς το παρόν κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος να παρεύει. Όχι. Ωραία. Ωραία λοιπόν περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι ένα άλλο θέμα για την ευθυγράμμιση. Η τροποποίηση του κανονισμού 485 του 2008 Συμβουλίου περί των ελέγχων εκ μέρους των κρατών μελών των ε, πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγύσεων. Εξηγητής είναι ο Λουίς Μανουέλ Καπούλα Σάντος, εξέταση του σχεδίου έκθεσης και εδώ η πρόταση αφορά μόνο τα θέματα ευθυγράμμισης. Λουίς, θες να παρέμβεις? Ευχαριστώ. Όπως είπε και η προηγούμενη συγκεντρία, μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα θέλουμε να καταργήσουμε το προηγούμενο σύστημα τη επιτροπολογία, αντικαθιστώντα το από το νέο σύστημα που έχει δύο επίπεδα τι εκτελεστικές πράξει και τι κατεξουσιοδότηση πράξεις θέματα που συζητούμε πια επανειλημμένω στην Επιτροπή μα. και μάλιστα έχουμε εκφράσει και αρκετέ ανησυχίε. Η δική μου πρόταση περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες τροπολογίες για να προσαρμοστούμε στη νέα κατάσταση και φυσικά με σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ο αποκλεισμό του κανονισμού από τα, με τα μέτρα ολοκληρωμένου ελέγχου και διαχείρισης που προβλέπουν ε, τα μέτρα για την ε, άμεση ενίσχυση. Προτείνει μια αναθεωρημένη εκδοχή επικαιροποιημένη του νομοθετικού κειμένου και προβλέπει τις προϋποθέσεις της εξουσιοδότησης προτείνουμε πενταετία και όχι χρόνο. χρόνου. Πενταετία που μπορεί όμως να παραταθεί αντίστοιχα κατά μία πενταετία αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και μάλιστα μέσα σε δύο μήνες μπορούν ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να εκφέρουν αντιρρήσει. και προτείνουμε τη διατήρηση ε, της Επιτροπής ε, του 1990 του 1995 σε σχέση με την Επιτροπή προτείνει ο δεύτερος κανονισμός. Αυτά και ευχαριστούμε τη Γραμματεία γιατί πρόκειται για ένα τεχνικό θέμα που είναι απαραίτητο για την προσαρμογή της συνθήκη της Λισαβόνας. Η Γραμματεία έδειξε και πάλι μεγάλο επαγγελματισμό και ικανότητα. Και για τις τροπολογίες διορία είναι και πάλι η 12η Απριλίου. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Λουίς. Πρόσωπο της Επιτροπής είναι η κυρία Μπουνιό. Ναι. Άρτη. Παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο. Η πρόταση της Επιτροπής όντως έχει στόχο την προσαρμογή του κανονισμού 485-2008 στη νέα νομική κατάσταση που δημιουργείται από τις ε, προβλέψεις της ε, ε, συνθήκης Λισαβόνας, άρθρα 2.90 και 2.91. Ε, πρόκειται μόνο για αυτή την ευθυγράμμιση, δεν προβλέπεται αλλαγή επί της ουσίας. Εμείς διαπιστώνουμε ε, με τεράστιο βαθμό σύγκλησης ανάμεσα στην πρόταση της Κομισιόν και το σχέδιο έκθεσης του κύριου Καπούλα Σάντος. Και ε, συμφωνούμε με τη διαχωρισμό μεταξύ των ε, κατεξοδότη πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων. Επίση, ε, στηρίζουμε την τροπολογία του κυρίου Καπούλα Άντε, που στόχο έχει την προσαρμογή στο κείμενο Common Understanding που πρόσφατα υιοθετήθηκε από τα τρία θεσμικά όργανα. Έχουμε μία ιδιαίτερη θέση αντίθετα όσον αφορά την τροπολογία 4 που είναι σχετική με την άσκηση των ε, κατεξοδότηση εξουσιών. Ο κ. Καπούλα Σάντο σας, προ... σας ε, εξήγησε ότι πρότεινε ε, ένα χρονικό περιορισμό για την παροχή των αρμοδιοτήτων στην Κομισιόν για, έξι για πέντε χρόνια. Η Κομισιόν προτιμά η υιοθέτηση των ε, κατοξιδότηση πράξεων να μην περιορίζεται χρονικά, να είναι επαόριστον και είναι μια πιθανή επιλογή μέσα στο πλαίσιο του Common Understanding. Η προσέγγιση αυτή νομίζουμε πως είναι πιο προσαρμοσμένη στις διτηρότητες της κοινή γεωργικής πολιτικής και στην ανάγκη άμεσης αντίδρασης η αποφυγής ε, μπλοκαρίσματος ε, και γνωρίζοντας βέβαια ότι σε κάθε στιγμή, ανα πάσα στιγμή η νομική αρχή μπορεί να άρει την εξουδότηση, να την καταργήσει. Έχουμε και ένα θέμα για την τροπολογία 3 που οι νομικοί μας ε, λένε ότι αυτή η τροπολογία, αν και είναι σωστή, δεν είναι απόλυτα απαραίτητη από νομικής άποψης. Αυτά, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Molto Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, κυρία Μπουνιό. Εφόσον δεν υπάρχουν παρεμβάσεις στο συναδέλφο, να δώσω εκ νέου το λόγο στο Λουίς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταγράφω ε, και σημειώνω με χαρά την μεγάλη σύγκληση που, υπάρχουμε, που υπάρχει με, εξέταση, με εξαίρεση το περιορισμό αυτών. Θα ήθελα να ξέρω την άποψη των συντονιστών των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Θα τους συμβουλευτώ και θα δούμε τελικά ποια στάση θα κρατήσουμε. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία ώστε να μπορέσει να περάσει αυτό το θέμα σε πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ. Οπότε τώρα ολοκληρώσαμε την εξέταση του σημείου 8. Θα κάνουμε 5 λεφτά διάλειμμα για να περάσουμε στο 9 και το ελαιόλαδο γιατί ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν έχει φτάσει ακόμα. Να σας ενημερώσω λοιπόν σε όλους τους κοσυντονιστές, παρόντες και απόντες, ε, στους απόντες μάλλον θα πρέπει να τους ε, ενημερώσετε γιατί μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση του σημείου του ελαιόλαδου που φαντάζομαι θα κρατήσει 20 λεπτάκια Αμέσω μετά θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Γι' αυτό θα έλεγα ότι μπορούμε να προβλέψουμε στις 5 τη συνεδρία των συντονιστών. Έτσι. Πέντε λεπτά διάλειμμα, περιμένουμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, να κάνουμε το τελευταίο σημείο, τα διάφορα δηλαδή, και μετά αμέσως η συνεδρία των συντονιστών.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 Έφτασε ο κύριος Φερστέλεν για να κλείσουμε με το τελευταίο σημείο στα διάφορα. Όπως είχα πει στην αρχή της συνεδρίασης, στη διάρκεια του τελευταίου Συμβουλίου Γεωργίας έγινε συζήτηση για την κρίση στον τομέα του ελαιόλαδου. Ε, αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές και μπορεί να είναι απαραίτητη η ιδιωτική αποθήκευση για να κάπως να διορθωθεί η κατάσταση. Ο Επίτροπος ε, Ντάσιαν Τσόλος υποσχέθηκε να λάβει υπόψη αυτή τη συζήτηση. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος που ο Διευθυντής Βερστάιλεν ήρθε και η Διαχειριστική Επιτροπή θα το συζητήσει νομίζω η επόμενη Διαχειριστική Επιτροπή στις 13 Απριλίου θα το συζητήσει, θα μας τα πει τώρα αυτά ο κύριος Διευθυντής. Νομίζω πως ή και η ώρα οι συνάδελφοι να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα του ελαιόλαδου. Αν και ο Επίτροπος είπε πολλές φορές ότι δεν πληρώνται οι ώρες για να ανοίξουμε στην ιδιωτική αποθήκευση, εγώ πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες που διανύει ο τομέας αυτός. Έγιναν διαδηλώσεις, ε, πολύ και στην Ισπανία, υπήρξαν προβλήματα στην Ιταλία. Ε, θέλουμε λοιπόν με κάποιο τρόπο να μπορέσει να δοθεί κάποιο μήνυμα προσοχής προς αυτό το τομέα που περνά μια περίοδο κρίση. Θα δώσω αμέσως το λόγο στους ε, βουλευτές που το ζήτησαν και μετά θα... Όχι, καλύτερα να ακούσουμε πρώτα τον Διευθυντή. Πρώτα τον κύριο Διευθυντή ε, για να μας ενημερώσει αν υπάρξει κάποιο νέο και μετά θα αρχίσει η συζήτηση και με τους ευρωβουλευτές. Το λόγο έχει αμέσως ο ε, κύριος Βερσλάιναν. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την εισαγωγή. Βεβαίω γνωρίζουμε την κατάσταση του ελαιολάδου στην κοινοτική αγορά. Ετέθηκε στο τελευταίο συμβούλιο το θέμα και ε, εκεί πέρα μας εξηγήθηκε πως για την ώρα στην Ελλάδα οι τιμές είναι κάτω του επίπεδου αν θέλετε στο οποίο θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ιδιωτική αποθεματοποίηση ενώ σε άλλες τιμές είναι πάνω από αυτό το επίπεδο και η νομική βάση λέει πως πρέπει να δείξουμε πως υπάρχει σοβαρή διαταραχή της αγοράς και ένα κριτήριο μετά είναι ε, το επίπεδο των τιμών. Και συμφωνούν πως οι τιμές είναι χαμηλές αλλά είναι πάνω από αυτό το επίπεδο παρέμβασης. Κατόπιν βεβαίως ε, συνεδρίασε η Διαχειριστική Επιτροπή του Συμβουλίου και το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Οπωσδήποτε βεβαίως τα κράτη-μέλη που είναι παραγωγή. Όλες οι πληροφορίες της αγοράς ε, που είχαμε διαθέσιμες, ε, που μας έστειλαν, για να έχουμε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και πως δεν υπήρχε διαφωνία στις τιμές, ποσότητες και τέτοια πράγματα και υπάρχει ακόμα αν θέλετε περιθώριο βελτίωσης και έναν παράγοντα μελετάμε ιδιαίτερα, δηλαδή το σε ποιο βαθμό σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη είχαμε μία πρώιμη σοδιά οπότε ίσως να υπάρχει περισσότερη διαθεσιμότητα αλλά αυτό είναι ένας παράγον που εξετάζεται ακόμα εξετάζουμε λοιπόν την κατάσταση και ε, από αυτή τη σκοπιά δεν μπορώ να πω εγώ τίποτα άλλο Ευχαριστώ. Eh, Μάλιστα. Δεν μας δώσατε και πολλές πληροφορίες, ούτε ελπίδες. Μήπως με τη συζήτησή μας μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Η Ράντς Γκαρσία ζήτησε το λόγο. Θα πρέπει να διαφωτίσουμε εμεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί φαίνεται ότι αγνοεί την κατάσταση στον τομέα. Εδώ και μία επταετία έχουμε σταδιακή μείωση των τιμών και μάλιστα τα τελευταία πέντε χρόνια είχαμε πραγματικά δραστική μείωση που είναι ανησυχητική για το τομέα και λόγω της παγκόσμιας μείωσης των τιμών, λόγω της άσκησης πίεσης εξαιτίας της χρήσης του ελαιόλαδου στη διαφήμιση για άλλα προϊόντα, λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής οι ελαιοπαραγωγοί χάνουν αγοραστική δύναμη με ε, άλματα και με ραχδαίο τρόπο. Ήδη το 2010 το μέσο κόστος παραγωγής ήταν 2,85 ευρώ και στην ε, Ισπανία λαμβάνουν 1,92 ευρώ. Βλέπετε τι τεράστια διαφορά υπάρχει μεταξύ της τιμής που λαμβάνουν και της τιμής κόστους, του κόστους της παραγωγής. Φανταστείτε σε τι ε, απόγνωση φτάνουν αυτές οι οικογένειες των ε, ελαιοπαραγωγών. Τι οικονομική κρίση αντιμετωπίζουν στις εκμεταλλεύσεις τους. Άλλωστε μιλάμε για ένα τομέα στον οποίο έχει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα τρίτο του παγκόσμιου ελαιολάδου παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 40% αυτού του συνόλου παράγεται στην Ισπανία και μάλιστα ιδιαίτερα στην Ανταλουσία. Εκεί το 25% του ΑΕΠ της Ανταλουσίας προέρχεται ακριβώς από τον τομέα παραγωγής ελαιολάδου. Οποιαδήποτε απόφαση λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει θεμελιώδη σημασία και τεράστιες επιρροές γιατί αφορά ένα εκατομμύριο ανθρώπους που εξαρτώνται άμεσα από τον τομέα ελαιολάδου στην Ισπανία μόνο να φανταστείτε ζητήθηκε η ενεργοποίηση του μηχανισμού ιδιωτικής αποθήκευσης, όπως έγινε τον Ιούλιο του 2009. Σήμερα συντρέχουν ίδιε προποθέσει με το 2009, για να μην πω ότι έχουν επιδεινωθεί όλα. Είναι λογικό να ενεργοποιηθεί αυτό ο μηχανισμό και μάλιστα όχι μόνο λογικό, είναι και απαραίτητο. Γιατί ούτε και οι μελλοντικέ προοπτικέ είναι ευίωνε με τη μεταρρύθμιση της κοινή ε, γεωρικής πολιτικής θα μειωθεί ακόμη περισσότερο η αγοραστική δύναμη των ελαιοπαραγωγών και θα μειωθούν τα εισοδήματά τους. Και μάλιστα, όπως σας είπα, δεν υφίσταται μόνο την πίεση των διανομέων, αλλά πλήττονται και από την έλλειψη νομικής ασφάλειας που χαρακτηρίζει το τομέα αυτό, που είναι πραγματικά σκανδαλώδης. Πριν από δύο χρόνια, ο ο τομέας αυτός προσπάθησε να οργανωθεί χωρίς να περιμένει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενεργοποιήσει την ιδιωτική αποθήκευση και να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Και μάλιστα έγινε και προσφυγή εναντίον τους, γι' αυτό και χρειάστηκε να διαλυθεί αυτή η οργάνωση. Και παρόλο που κέρδισαν μετά στο κυρωτικό δικαστήριο, δεν είχαν πια χρήματα για να επανανεργοποιήσουν αυτόν τον μηχανισμό. Προσπάθησαν να διασωθούν, αλλά Δυστυχώ ε, δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν αυτό το μηχανισμό. Και τώρα που νομικά υπάρχει δυνατότητα να το κάνουν, δεν έχουν πια την οικονομική ε, δυνατότητα. Δεν υπάρχει καν νομική ασφάλεια δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να ενεργούν ε, ε, με παρόμοιε συνθήκε όπω και άλλοι τομεί. Φυσικά θέλουμε ενεργοποίηση της ιδιωτικής, ε, της, του μηχανισμού αποθήκευση. Οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν να ενεργοποιήσουν και μηχανισμό ιδιωτική αποθήκευση για να άρουν κάπως τα αρνητικά αποτελέσματα τη ανασφάλεια δικαίου που επικρατεί στον τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την Παρασκευή που θα πραγματοποιήσει και η επίσκεψη ο Επίτροπος Γεωργία στην Ισπανία να επιτραπεί η ενεργοποίηση της ιδιωτικής ε, αποθεματοποίησης που είναι απαραίτητη και εν ώψη της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει και να προτείνει μηχανισμούς για να σωθούν περιοχές ε, με το νέο σύστημα της ε, βοήθειας αναεκτάριο, της ενίσχυσης αναεκτάριο, γιατί η, επίδραση αυτής της, η συνέπεια αυτής της πρότασης μπορεί να οδηγήσει στην Ανταλουσία και στην απώλεια του μισού του σχεδόν εισοδήματος, του 50%. Δεδομένη στις αρνητικές κατάστασεις που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια, θα είναι τραγική μια τέτοια εξέλιξη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, κυρία Χεράντ Γκαρσία. Ζήτησε το λόγο και ο κύριο Άγνιου. Και μετά θα πω και εγώ δύο λόγια. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με ενδιαφέρον βλέπω, ε, βεβαίω δεν παράγω και κανείς στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν παράγει ελαιόλαδο, βλέπουμε πως ε, μπορεί να αλλάξει, να είναι... Το λάδι από ελαιοκράμβη είναι εναλλάξιμο με το ελαιόλαδο και ξέρετε πως έχει πάει από τους 200 λίρες στις 400 λίρες τον τόνο η τιμή του. Οπότε είναι ενδιαφέρουσα η σύγκριση και αναρωτιέμαι εάν η Κομισιόν μπορεί να σχολιάσει αυτή την ε, αντίφαση. Επίσης θα ήθελα να μου πούν αν έχουν κάνει κάποια έρευνα για τις λιανικές τιμές. Τουλάχιστον επωφελείται ο καταναλωτής από τη μείωση τιμών παραγωγού ή κάποιος ενδιάμεσος ε, κερδίζει πολλά χρήματα. Ευχαριστώ, Λουίς έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να ενισχύσω και να στηρίξω την παρέμβαση της συναδέλφου Έρανς Γκαρσία γιατί είναι ένα πραγματικό πρόβλημα και όταν εμεί συζητάμε την κοινή γεωργική πολιτική και επιμένουμε για την ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών ρύθμισης αγοράς δεν μιλάμε για αόριστα πράγματα, μιλάμε για μηχανισμούς που πρέπει να είναι λογικοί για να λύνουν τα προβλήματα όταν η αγορά δεν καταφέρει να δώσει απάντηση με την ε, λειτουργία της. <coughs> και αυτή είναι μια περίπτωση προφανής νομίζω. Γιατί αντίθετα με όλες τις προβλέψεις σε σχέση με την αύξηση κατανάλωση κατανάλωσης ε, παγκοσμίω που είχαμε διαβάσει τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνουμε πως ε, τιμές μειώνονται σταδιακά και ότι ε, από πλευρά τη Κομισιόν υπάρχει μια υπερβολική, ένας υπερβολικός δισταγμός για ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα σε πολλά κράτη-μέλη. Και γι' αυτό ήθελα να δώσω έμφαση στην ανάγκη να αντιδράσει γρήγορα η Κομισιόν με τα, τους μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή της. Και νομίζω πως αυτό που άμεσα μπορεί να χρησιμοποιήσει είναι η ιδιωτική αποθήκευση για να δοθούν απαντήσεις σύντομα. Ευχαριστώ, Λουίς. Ο κύριος Γιάρας έτσι το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, και εγώ δεν είμαι κανένα ειδικό ε, για τον κανονισμό του ελαιολάδου, αλλά ο Άγγλος συνάδελφος με ενθάρρυνε και με να ρωτήσω, γιατί δεν μας διαφώτισε η Κομισιόν και ήταν πολύ σύντομα αυτά τα οποία είπε. Οπότε το ερώτημά μου είναι Ποια θεωρεί η Κομισιόν την αιτία για τις χαμηλές τιμές. Υπάρχει μεγάλη παραγωγή στην Ευρώπη, ωφελείται στην παγκόσμια αγορά. Ή κάπου στην αλυσίδα κάποιος βγάζει υπερκέρδη. Και αν ε, υπάρχει κάποιες, αν έχει κάποιες αναλλακτικές ε, να προτείνει η Κομισιόν για να βελτιωθεί η τιμή του καταναλωτή. Και τέλος, ε, προς την συνάδελφο, Όταν μιλάμε για το μέσο παρέμβαση στην αγορά, το ερώτημά μου είναι ε, ποια ποσότητα ε, σκέφτεται η Κομισιόν και για πόσο χρόνο θεωρείται ότι πρέπει να παρέμβει και βέβαια με ποιο σκοπό. Μάλιστα και εγώ θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρέμβαση δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να θέλουν να πάρουν το λόγο και θα απευθύνω και εγώ μια ερώτηση στον ε, κύριο Φερστάιλιν. Σίγουρα δεν ε, έχετε φτάσει, είπατε, στο επίπεδο του ελάχιστου το ελάχιστο κατόφλι που επιτρέπει την λήψη επιγόντων μέτρων. Μήπω όμω θα πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε, να αναθεωρήσουμε αυτό το μηχανισμό που ορίζει το κατώτερο κατόφλι, γιατί δεν είναι δυνατόν ενώπιον μια σαν ευπροηγουμένου κρίση στην Ισπανία, στην Ιταλία και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Άμα δεν λειτουργεί, θα πρέπει ίσω να αλλάξουμε το μηχανισμό ώστε να λειτουργήσει. Εμεί έχουμε και κάποια νομοθετικά πακέτα υποσυζήτηση. Έχουμε νομοθετικά μέσα που θα μα επέτρεπαν να το κάνουμε αυτό, αν συμφωνεί η και Δεύτερο ερώτημα. Ε, δεδομένου ότι για την ε, ΚΟΑ, για τα ποροκυπευτικά, στην τελευταία μεταρρύθμιση που κάναμε το 2007, φτιάξαμε μηχανισμούς διαχείρισης κρίσης που φαίνεται να λειτουργούν πολύ καλά στη διαχείριση της κρίσης, ε, που... μηχανισμούς που εισάγαμε στην τελευταία μεταρρύθμιση. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν και στο τομέα του ελαιολάδου να εισάγουμε αντίστοιχους μηχανισμούς για να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να διαχειρίζονται καλύτερα την προσφορά στην αγορά. Τα τριετή προγράμματα αυτή τη στιγμή λειτουργούν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν επέτρεψαν πολλές βελτιώσεις από την άποψη της ομαδοποίησης, της προσφοράς και της διαχείρισης της κρίσης. Και εδώ λοιπόν μια ερώτηση. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια φάση εντατική νομοθετικής παραγωγής, μήπως θα ήταν σκόπιμο τόσο για τον καθορισμό της τιμής του κατώτερου ορίου ο καθορισμό δηλαδή μια τιμή που να λαμβάνει υπόψη ένα μήνυμο ευελιξία για τα κράτη. Και έπειτα, όσον αφορά αντίστοιχα μέσα, όπως το πρότυπο τη ε, ΚΟΑ για τα προκυπτικά. Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη σε επίπεδο κομισιών. Αυτές είναι οι ερωτήσει που ήθελα να κάνω και θα ήθελα να δώσω το λόγο εκ νέου, εάν δεν υπάρχουν συνάδελφοι που να θέλουν να παρέμβουν εντωμεταξύ. μεταξύ στον κύριο Διευθυντή για να μας ε, απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις με τη σειρά που τέθηκαν. Η κυρία Ράνς Γκαρσία αναφέρθηκε σε πιθανή μείωση της ενίσχυσης ανά εκτάριο. Γνωρίζουμε ότι αυτή η ενίσχυση είναι σημαντική όχι μόνο στο τομέα παραγωγή, αλλά και σε άλλου τομεί. Αλλά από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει καμία πρόθεση μείωση τη ενίσχυση στο ελαιόλαδο. Ενίσχυση σαν εκτάριο δηλαδή. Αλλά θα αποτελέσει τμήμα τη γενικότερη συζήτηση για το μέλλον τη κοινή γεωρική πολιτική μετά το 2013 και το κατά πόσο θα παραμείνει αυτό το σύστημα ενίσχυση σαν εκτάριο αλλά δεν θα είναι ένα ειδικό μέτρο για το ελαιόλαδο αυτή η μείωση της ενίσχυση ανακτάριου. Θα είναι κάτι γενικό αν συζητηθεί. Σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση Ελαιόλαδο από, ελαιο, από ελαιο, Σε μερικές περιπτώσεις ε, γίνεται τέτοια αντικατάσταση, είτε στο μαγείρεμα ή σε πολλές χώρες το κάνουν. Αλλά τώρα η σε πολλες χώρε το σχέση ελαιόλαδου και ελαιοελαιοκράμβη δεν νομίζω ότι είναι απολύτως αντίστοιχα. Και υπάρχει και θέμα συγκυρίας για το ελαιόλαδο. Συνήθως όταν υπάρχει μεγάλη προσφορά ελαιολάδου γίνεται σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου. Είχαμε 420.000 τόνου τόνους στην Ισπανία αρχικά, αλλά και μια και φέτος η εισοδιά ήταν λίγο νωρίτερα έχουμε 1,1 εκατομμύριο τόνους. Και αυτό φυσικά έχει επιρροή στην αγορά αυτή η αύξηση της παραγωγής και εξηγεί έτσι και τις χαμηλές τιμές. Τώρα, στο, σε ποιο βαθμό αποφελείται και ο καταναλωτής από τη μείωση των τιμών, αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι όντως αποφελείται και ο καταναλωτής, γιατί Ήδη υπάρχουν κάποιες δράσεις σε ελοπαραγωγές χώρες, γιατί τα σούπερ μάρκετ χρησιμοποιούν ε, το ελαιόλαδο ως ε, τρόπο διαφήμισης ε, και προβάλλουν, ας πούμε, τη χρήση του ελαιολάδου στις σαλάτες. Για παράδειγμα, στο βορρά προβάλλεται ιδιαίτερα η χρήση του γάλακτος. Στο νότο προβάλλεται περισσότερη χρήση του ελαιολάδου. Και κάτι τέτοιο φυσικά επηρεάζει τις τιμές γιατί τα σούπερ μάρκετ ενδιαφέρονται να καρποθούν ένα μεγάλο τμήμα φυσικά αυτής της διαφοράς. Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση που επισήμανε ο κύριος Καπόλα Σάντος και το επίπεδο δικτύου ασφαλείας για το ελαιόλαδο. Αυτή ήταν η τιμή, αναφορά, αναφοράς, αυτό το safety net level, και με αυτή τη τιμή αναφοράς, ε, με αυτό το κατόφλι ενεργοποιείται η ιδιωτική αποθεματοποίηση, εφόσον συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις. Αλλά δεν έχουμε μόνο το, την τιμή ως αξία για την ενεργοποίηση. Υπάρχει ένα περιθώριο λιγμών και διακριτική ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη και την ε, συγκυριακή κατάσταση και το κατά πόσο θα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό της ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Δεν είναι μόνο η τιμή λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις ε, του κ. Κάστρο, του Πρόεδρου, αν το επίπεδο της τιμής αναφοράς είναι προσαρμοσμένο στη σημερινή κατάσταση. Και εδώ σα παραπέμπω στην ευρύτερη συζήτηση που γίνεται για το safety net, για το δίκτυο ασφαλεία και το κατόφλι ενεργοποίηση του μηχανισμού. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το ελαιόλαδο, αλλά και για άλλου τομεί. Έχουμε καταλήξει έμεσα στο συμπέρασμα ότι θεωρούμε το επίπεδο ενεργοποίηση επαρκέ για του περισσότερου τομεί. Αλλά μετά το 2013 που θα συζητηθεί, με θα ισχύσει η νέα ΚΑΠ, θα, το, θα δούμε αν θα διατηρηθεί αυτό το κατόφλι ή θα τροποποιηθεί. Δεν ξέρω, έχω κάποιες αμφιβολίες, πάντως ε, είναι τμήμα της γενικότερης συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Και σε ό,τι αφορά την τελευταία σας συζήτηση για παρα, αντίστοιχα παραδείγματα στα απορροκυπευτικά, η ιδέα αυτού, αυτών των ομάδων ε, παραγωγών και της ε, εξουσίας διαπραγμάτευσης θα μπορούσα να σκεφτώ και αυτό το στοιχείο, γιατί είναι σημαντικό και για τον, τον κλάδο του ελαιολάδου. Δηλαδή, οι ασθενείς θέσει της, των Ισπανών παραγωγών απέναντι στους διανομείς θα πρέπει να εξεταστεί γιατί το, και θα πω σε σκοπιμότερο να οργανωθούν καλύτερα μεταξύ τους για να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους ε, δύναμη απέναντι στους, ε, στις μεγάλες αλυσίδες διανομής. Αλλά και αυτό θα, θα εξεταστεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ μετά το 2013. Σα ευχαριστώ που μα δώσατε κάποιο τελικό άνοιγμα. Οπότε καλώ του συναδέλφου, Εράν Γκαρσία, Λουίς Κάπολα, Σάντος και όλου του συναδέλφου που είναι πιο κοντά στην μεσογειακή παραγωγή να σκεφτούν μήπω θα ήταν σκόπιμο να δεχτούμε την πρόσκληση του κυρίου Διευθυντή, να σκεφτούμε το πακέτο γάλακτο για να ε, επεκτείνουμε και κάποιου μηχανισμού διαχείριση τη κρίσης. Σα ευχαριστώ τέλο τη συνεδρία, σα Θυμίζω τι ημερομηνίε για την επόμενη συνεδρία, 11 Απριλίου στι 3 και 12 Απριλίου στις 9. Ευχαριστώ όλους. Τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής και ξεκινάει η συνεδρία των συντονιστών.